Θέλει να πάρει το λόγο η εισηγήτρια πριν την ψηφοφορία. Ναι, συντομία, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω καταρχά όλου του κοιότε εισηγητέ. Η συνεργασία του ε, αυτή την πολύ δυτική περίοδο ήταν πραγματικά κρίσιμη για να πετύχουμε προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και καταφέραμε να αυξήσουμε την εντολή μια τόσο σημαντική υπηρεσία. Η υπηρεσία αυτή λοιπόν θα φτάσει τις 10.000 θέσει μέχρι το 2027 και θα είμαστε σε καλύτερη θέση να βοηθήσουμε τα κρατημέλη σε ό,τι αφορά τι επιστροφέ και όλε οι θέσει αυτέ έχουν να κάνουν με θεμελιώδη δικαιώματα. Το κείμενο περιλαμβάνει και πιο ισχυρέ υποχρεώσει σε ό,τι αφορά την υποβολή αναφορών προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώ και πιο ξεκάθαρη διατύπωση για το πότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καλείται να συμμετέχει σε συνελεύσει του Διοικητικού Συμβουλίου. Μία επιπλέον σημείωση, σημαντική θεωρώ, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν επί μια κοινή δήλωση και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την αμοιβή του προσωπικού της υπηρεσίας. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και την αναθεώρηση του κανονισμού των Ευρωπαίων υπαλλήλων, προκειμένου να εξασφαλίσουμε και πάλι ότι η Frontex θα είναι μια ελκυστική υπηρεσία για να εργάζεται κανείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία, ιδιαίτερα στην Κάθριν και τον Γιάννη και καταφέραμε, θεωρώ, να διαπραγματευτούμε ένα κείμενο το οποίο συνάδει με την εντολή που έλαβα από την Επιτροπή μας και ελπίζω να μπορέσουμε να αποστείλουμε ένα καλό και γύρω μήνυμα προς όφελος της υπηρεσίας από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λέκη Πρόεδρος. Και να περάσουμε στις πληροφορίε για το κείμενο που συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια των διαθεσμικών διαπραγματεύσεων. Έναρξη της ψηφοφορία. Ψήφισατε παρακαλώ όλοι. Έχουμε δύο υπεράριθμους από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Έναν ακόμα. Μάλιστα. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η ψηφοφορία και από σοσιαλδημοκράτες περισσεύει Σε Ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Μακάρι να θέλουν να ψηφίσουν όλοι έτσι και στα δικά μου τα θέματα. Αλλά τα δικά μου θέματα δεν έχουν να κάνουν με ασφάλεια. Πέρα ψηφοφορία τώρα. 33 ψήφοι υπέρ, 13 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. So, um, so we have a, um, there is another vote. Άλλη μια ψηφοφορία. Συνάδελφοι, έχουμε ακόμα μία ψηφοφορία. Πού πάτε? Έχουμε άλλη μία ψηφοφορία, λέω. Όχι. Okay. Okay, sorry, colleagues. Just... συγγνώμη, συνάδελφοι. Σας παρακαλώ να δείξετε υπομονή. Καθίστε λίγο ακόμα. Δεν σας έχουμε ενημερώσει να σας εξηγήσω ότι έχουμε την ψηφοφορία Σας παρακαλώ συνάδελφοι, ακούστε με λίγο. Ένα λεπτάκι. Κάντε λίγο υπομονή στα πίσω έντρανα. Έχουμε λοιπόν το θέμα των τρίτων χωρών και τι θεωρήσεις σε ό,τι αφορά τι σχετικέ προδιαγραφέ, σε ό,τι αφορά και την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έλαβε χώρα ένα τριμερή διάλογο με το πρωί με τον νέο, με τον εισηγητή, τον κ. Στάνισλεφ, και ε, λάβαμε μόλι ε, νέα ότι επιτευχθεί μια συμφωνία σε ό,τι αφορά. Σας παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Κάντε λίγη ησυχία. Και η σύγχυση που έχει προκληθεί με οδηγεί στην εξή απόφαση. Λάβαμε λοιπόν την επιστολή από την Κορεπέρ που επιβεβαιώνει τη συμφωνία και μπορούμε να κάνουμε την ψηφοφορία. Σας παρακαλώ, αφήστε με να τελειώσω. Προφανώς όμως πολλοί από εσά δεν έχετε υπόψη σας τι έχει συμβεί. Άρα είτε θα ψηφίσουμε τώρα είτε εναλλακτικά και επιτρέψτε μου το ελέγξω με τη γραμματεία. Μπορούμε να ψηφίσουμε αύριο στις 8.30 το πρωί. Yeah, just one second. Okay. Μισό λεπτό, λέει ο Πρόεδρος. Μισό λεπτό. Δώστε μου μισό λεπτό. Δεν είμαι υπεύθυνο εγώ για το θέμα αυτό, για το φάκελο αυτό και δεν είμαι εγώ αυτό που ευθύνομαι για το χάο που επικρατεί. Να σα εξηγήσω μισό λεπτό ποιε είναι οι εναλλακτικέ. Καταρχά. Μ' ακούτε? Έφτασε λοιπόν η επιστολή από την Κορεπέρ. Ο εισηγητή δεν είναι εδώ. Θα καταφτάσει στι 4.30. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πρόβλημα. Αν έχετε οποιοδήποτε θέμα λοιπόν αναφορικά με την έκθεση, δεν είναι εδώ ακόμα. Θα έρθει στι 4.30. Θα είναι και εδώ αύριο στι 8.30, αν η ψηφοφορία λάβει η χώρα αύριο το πρωί. δεν είναι όμω τώρα εδώ. Αν όλε οι ομάδε, όλε οι ομάδες επαναλαμβάνω, επειδή είναι ευαίσθητο το θέμα, θέλουν να ψηφίσουν τώρα, γιατί του βολεύει καλύτερα, μπορούμε. Εναλλακτικά μπορούμε να ψηφίσουμε αύριο το πρωί στις 8.30 το πρωί και θα έχουμε στη διαθέσή μας και τον εισηγητή. Υπάρχουν άλλες επιλογές? Όχι. Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Αυτές είναι οι εναλλακτικέ που έχουμε στη διαθέσή μας. Και δεν φταίω εγώ. Δεν είναι δικό μου ο φάκελος. What do you want to do? Τι θέλετε να κάνουμε λοιπόν για το θέμα του κυρίου Στάνισλεφ για τις θεωρήσεις. Κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και το τσακάρισα. Ο Σέρκεϊ, ο νέος εισηγητής, ζήτησε να γίνει ψηφοφορία αύριο το πρωί, γιατί αυτός ήταν που ολοκλήρωσε το φάκελο και ήθελε να είναι παρόν. Επίσης θα ήθελε να δώσει σε όλους και λίγο χρόνο να το σκεφτούν προτού πάρουμε μια βιαστική απόφαση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσουν να γίνει ψηφοφορία αύριο το πρωί. Ο Πρόεδρος. Άλλος κανείς. Κοιτάξτε, μην ακούω μόνο μουρμουριτά. Θέλω μόνο προτάσεις να ακούσω υπέρ κατά όπως αυτή της κυρίας Σίπελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι ευαίσθητο θέμα αυτό για το Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ δεν είμαι προετοιμασμένο για να προχωρήσω σε ψηφοφορία τώρα. Μου είχαν πει ότι θα υπήρχε αναβολή αύριο το πρωί στις 8.30 και μιλάτε εξ ονόματος του EFTD, όχι του ENF. Του ENF και εσεί, ε, κύριε Ζήλστρα, Σοσιαλιστέ και δημοκράτε και η ΕΝΕΦ. Ενδιαφέρον ο συνδυασμό. ECR. Ε να ακούσουμε μια άποψη του το ECR. Ε ναι, κοιτάξτε, από δικέ μα πλευρά και εγώ να πω ότι χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω χρόνο να εξετάσουμε τι λεπτομέρειε τη τελική συμφωνία. Άρα θα προτιμούσα να ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Ησυχία, ναι. Άλτε σας ευχαριστώ ως συντονίστρια της Άλτα. Θέλουμε να είναι παρόν και εισηγητής, να σεβαστούμε την ε, αξίωση του να είναι και αυτός παρόν κατά τη διάρκεια της ψηφορίας, άρα 8.30 αύριο το πρωί. Μάλιστα. Έχω την εντύπωση ότι δεν ε, προτιμάτε να γίνει τώρα η ψηφοφορία. Είναι κανείς που είναι αντίθετος με την ψηφοφορία αύριο στις 8.30? Όχι. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε άλλη μία ψηφοφορία αύριο το πρωί στις 8.30 με παρουσία του εισηγητή. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες σήμερα.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 δεν ε, μπορώ να πω αν είστε δανός έτσι εξόψεως. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. But you're welcome up here. Αλλά είστε πρόσδεκτοι εδώ, στο βήμα. And anyone who's staying for this, uh, staying for this point, please. Παρακαλώ, όποιος θέλει να παραμείνει για αυτό το σημείο, να καθίσει. Okay, colleagues, the next Το επόμενο θέμα είναι η απόφαση του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τη συμφωνία Eurojust και Δανία. Συμφωνήσαμε χτες. Συμφωνήσαμε ότι θα σημειώσουμε πρόοδο για το θέμα αυτό. Στη κανονισμός του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της του Νεμβρίου του 2018 για τη Eurojust ε, υιοθετήθηκε και καταργήθηκε η απόφαση του Συμβουλίου η σχετική και ε, λησβονοποιήθηκε, λησβονοποιήθηκε η Eurojust ε, από το Δεκέμβριο του 2019 κτλ του 2018, συγγνώμη. Η Δανία λοιπόν δεν συμμετέχει στο νέο κανονισμό, δεν δεσμεύεται από αυτό. Παρ' όλα αυτά η Δανία έχει εκφράσει την επιθυμία να συμμετέχει περαιτέρω στις δραστηριότητες Eurojust. Έτσι λοιπόν η συμφωνία συνεργασίας πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ Eurojust και Δανίας, παρόμοια με τη συμφωνία την οποία ε, είχε συνάψει με τη Europol η Δανία. Έτσι λοιπόν, είχαμε μια, ένα σχέδιο απόφαση συμβουλίου που εθετήθηκε στο Γιουροπέρ και την 1η Απριλίου εστάλει στο Κοινοβούλιο για έγκριση. Τρει μήνε είναι η συνήθιση προθεσμία. Υπό τη διαδικασία αυτή, το Κοινοβούλιο μπορεί να εγκρίνει, να μην εγκρίνει το σχέδιο απόφαση συμβουλίου μέχρι μια συγκεκριμένη προθεσμία. Δεν μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο τη εφαρμοστική συμφωνία. Η Δανία έχει εκφράσει την επιθυμία να ολοκληρώσει τη συμφωνία το συντομότερο και να υπάρξει ταχεία δράση του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Ε, και η Επιτροπή θα ξεκινήσει τη διαδικασία και θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει εντό αυτή τη θεία. Προτείνω το εξή χρονοδιάγραμμα. Σήμερα, 2 Απριλίου, να παρουσιάσουμε το σχέδιο συμφωνία. Αυτό κάνουμε τώρα στι 8 Απριλίου. Θα ψηφίσουμε στη Λίμπε και κατόπιν ε, θα ψηφίσουμε στην ε, δεύτερη ολομέλεια του Απριλίου. Η απλουστευμένη διαδικασία είναι μόνο στα αγγλικά, χωρίς τροπολογίες. Δεν υπάρχουν υποσημείωση τροπολογίες, παρακαλώ. Και ιδίω επειδή θα είμαι ο πρόεδρος. Και θα προσπαθήσουμε να το ψηφίσουμε στη δεύτερη σύνοδο του Απριλίου. Και επειδή η Δανία το έχει κάνει δύο φορές, ε, δεν θέλω ομπελάδες. Σας προειδοποιώ, θα δώσω τώρα το λόγο στη Eurojust στην Προεδρία, στην Κομισιόν. Έτσι λοιπόν και στους εκπροσώπους της Δανίας ε, κάνουμε κάτι καλό για σας. Thank you very much. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και που εφαρμόζετε αυτή τη ε, διαδικασία, η συμφωνία αυτή αφορά τη Europest. Κοιτάξτε, η Προεδρία και το Συμβούλιο έχουν ε, συμβάλει. Όπως και να έχει, σας ευχαριστούμε. Γιατί, τι θέλουμε να κάνουμε να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουν οι εργασίες με τη Δανία. Έχουμε 252 υποθέσεις που συνεχίζονται με τους δανούς συναδέλφους στη Eurojust, που υποστήριζονται από τη Eurojust και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το έργο στο μέλλον. Σας έχουμε στείλει κάποια στατιστικά στοιχεία. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Δανία έχει μεταξύ 4,5 και 7,5% όλων των υποθέσεων στη Eurojust. Έτσι λοιπόν δεν μιλάμε για μινιμαλιστικές ε, υποθέσεις, αλλά πολύ σοβαρές και σημαντικές υποθέσεις, ε, όπως ε, την περίπτωση της τράπεζας Danske ή επιχειρησιακός οργανισμός. Όλα αυτά έχουν ως σκοπό να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τη Δανία. Έχουμε εμπνευστεί από το εφιστάμενο κανονισμό η πρότυπη συμφωνία Eurojust με τα τρίτα κράτη γιατί ουσιαστικά γίνεται λειτουργικά τρίτο κράτος η Δανία αλλά θα παραμείνει κράτος μέλος. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να γίνει προσαρμογή. Έχουμε και τη συμφωνία Δανίας Europol του 2017 αλλά Κατόπιν αυτού είχαμε νέους κανόνες για την προστασία των δεδομένων που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Φυσικά ο κανονισμό Eurojust του 2018 και έχουμε και την οδηγία περί του 2016. Τι θέλουμε να κάνουμε τώρα σε σύγκριση με τα τρίτα κράτη. Να δώσουμε στη Δανία ένα ειδικό καθεστώς στη Eurojust. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι παρατηρητές στο σώμα μας και θα έχουμε τον δανό εκπρόσωπο και όχι τον αξιωματικό δικαστικό σύνδεσμο, όπως ε, τους αποκαλούμε τώρα. Θα έχουμε δημοκρατική εποπτεία από το Δανέζικο Κοινοβούλιο και θα λαμβάνουν μία αιτήσια έκθεση για το τι έχουμε κάνει, αυτό που κάναμε πάνω κάτω σήμερα το πρωί, και θα έχουμε και τη δυνατότητα απόσπασης ενός ε, ε, ε γραφείου εκπροσώπων για τη Δανία. Επίσης, ε, θα υπάρχουν ειδικές, ειδικά δικαιώματα και ειδικέ υποχρεώσεις και έχουμε και την οικονομική συνεισφορά που θα καταβάλει η Δανία, όπως έχουμε και στη συμφωνία με την Europol, έχουμε και τον περιορισμό του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου και την εποπτεία του Ευρωπαίου Επόπτη για την προστασία των δεδομένων. Αυτά όλα τα έχει αποδεκτεί η Δανία και τα καλωσορίζει. Παράλληλα, έχουμε ελέγξει το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Έχουμε αξιολόγηση από το αρμόδιο όργανο προστασίας των δεδομένων και μας είπε ότι είναι εύρωστο και σύγχρονο το σύστημα και συμπεριλαμβάνει όλους τους νέους κανόνες, ιδίως το δεσμευτικό κανόνα της ε, οδηγίας για την αστυνομία για τη Δανία. Και φυσικά υπάρχουν και όλοι οι κανόνες ε, που θα ισχύουν και στο νέο κανονισμό. Συνολικά νομίζω ότι είναι εφικτό και γρήγορο το σύστημα και θα μπορούσαμε εύκολα να το εφαρμόσουμε όταν ε, θα αρχίσει να ισχύει ο νέος κανονισμός γύρω σας στις 12 Δεκεμβρίου 2019 και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ταχεία διαδικασία για να πετύχουμε ταυτόχρονα ε, να συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Μάλλον ε, έπρεπε να δείξουμε και αυτές τις διαφάνειες με την ομιλία σας. Τέλο πάντων, αστείευομαι. Λοιπόν, Προεδρία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί σχεδόν όλα υπόθηκαν από τον κλάου τον Αντιπρόεδρο τη Eurojust. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ και τη Eurojust και τη Δανία που κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντική στιγμή για το Συμβούλιο και εντό του Συμβουλίου υποστηρίξαμε πλήρως ταχείες διαπραγματεύσεις και ταχεία θέτηση αυτής της συμφωνίας γιατί πιστεύουμε ότι δεν εξυπηρετεί μόνο το συμφέρον της Δανίας και της Eurojust, αλλά είναι και σημαντική για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, είναι η καλύτερη δυνατή λύση υπό αυτές τις συνθήκες, καθώς η Δανία δεν μπορεί να ξεκινήσει στις 12 Δεκεμβρίου ως, πλήρως μέλος, ως πλήρες μέλος της Eurojust. Αλλά πιστεύουμε ότι η Συμφωνία για την συνεργασία σε δικαστικές ποινικές υποθέσεις είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση. Καθώς ουσιαστικά η Δανία θα έχει μια ειδική σχέση με τη Eurojust. Φυσικά από τη σκοπιά του κανονισμού θα τύχει μεταχείριση τρίτης χώρας, αλλά καθώς είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κράτος μέλος, δικαιολογείται να έχει αυτό το ειδικό καθεστώ. Και δεν είναι ότι το αξίζει πλήρω ε, η Δανία απλώ. Δεδομένου ότι την ε, σημαντική συνεισφορά της στην ανάπτυξη της Eurojust τα τελευταία 17 χρόνια ως ε, ιδρυτικό κράτος μέλος της Eurojust. Αλλά, όπως είπα, είναι και προς το συμφέρον της Ένωσης να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό θα ήταν δυνατό μόνο με μια τέτοια συμφωνία. Για να διατηρηθεί η σημερινή συνεργασία, όχι μόνο μεταξύ Δανίας και Eurojust, αλλά και μεταξύ όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στη Eurojust. Και καταληκτικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δέχτηκε να γνωμοδοτήσει υπό σημερινή θητεία. Είναι σημαντικό και συμφωνήσαμε όλοι στο Συμβούλιο η συμφωνία αυτή να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο. Και πιστεύουμε τώρα ότι είναι δυνατόν να υιοθετηθεί εντός της δικής μας Προεδρίας του Συμβουλίου, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε οποιοδήποτε επιχειρησιακό κενό που μπορεί να προκύψει. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι από τις 12 Δεκεμβρίου η Δανία θα μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες της Eurojust σχεδόν σαν πλήρες μέλος, όπως εξήγησε ο Κλάους, μέσω των εκπροσώπων της. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία στη Δανία και στη Eurojust για τη μελλοντική του συνεργασία υπό το νεονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όντω ήταν η... η δεύτερη καλύτερη λύση. Η καλύτερη θα ήταν να έχει παραμείνει ω πλήρε μέλο τη Eurojust στη Δανία. Αλλά μια και υπάρχει ειδικό καθεστώ και δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή. Η συμφωνία για το μοντέλο της συμφωνίας Europol-Δανίας είναι η δεύτερη καλύτερη, όπως είπα και είπαν και οι προλαλήσαντες, ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, ομαδική δουλειά που αναπτύξαμε η ομάδα της ε, Europol ε, που να παρούσα, η Δανική κυβέρνηση, η Επιτροπή έτσι ώστε να τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις για τη λειτουργική συνεργασία με καθεστώς προστασίας που πρέπει να ισχύει και για τη Δανία ε, υπό τους όρους της Οδηγίας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Άρα υποστηρίζουμε πλήρως τη συμφωνία. Για διάφορους λόγους επιτρέψαμε να εκθέσω μερικούς εξ αυτών. Καταρχάς γιατί είναι προς το συμφέρον των πλευρών της Eurojust και της Δανίας, η ολοκλήρωση τη Συμφωνία, η σύναψη της συμφωνίας, ώστε να παραμείνει μέσα στην οικογένεια της Eurojust στη Δανία. Θα έχει τη δυνατότητα να συνεδριάζει στις, στις συντονιστικές ε, αλλά και στις στρατηγικέ στρατηγικές ε, συνεδριάσεις. Άρα θα έχει περισσότερη συμμετοχή από ότι μια οποιαδήποτε τρίτη χώρα έναντι της Eurojust. Επίσης η Δανία συμμετέχει σε διάφορες συμφωνίες ε, τρίτου πυλώνα νομοθετικές πράξεις όπως το Ευρωπαϊκό Ένταλμα για διάθεση Αγράφων και άρα θα βελτιωθεί η συνεργασία της τρίτων. Είναι μέλος της Σέγγεν Δανία. Και άρα συμμετέχει σε μια σειρά από δραστηριότητες. Με την Έτσι λοιπόν το να παραμείνει μέσα στην Eurojust είναι πολύ το σημαντικό εδώ. Πρέπει να εξασφαλίσουμε και ένα πεδίο ισότιμο για τη Δανία, ώστε και η αστυνομία της να μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες της Europol και άρα σε αυτό πρέπει να ενσωματωθεί και η διάσταση των ε, διοκτικών αρχών. Επίσης για το Εθνικό Κοινοβούλιο έχει πολύ μεγάλη σημασία είδαμε και τις αιτήσει εκθέσεις της Eurojust. Ο δικαστικός έλεγχος που προβλέπεται στη συμφωνία είναι ευπρόσδεκτος. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα εξετάσει τις διατάξεις ε, για να τις ερμηνεύσει αν χρειαστεί. Και βέβαια στο θέμα του κανονισμού η την προσέγγιση προσωπικών δεδομένων θα υπάρχει σχετική επαλήθευση. Εν τέλει και πολύ σημαντικό, η Δανία συμμετέχει και στον προϋπολογισμό της Eurostat με βάση μια κλίδα που προβλέπεται στο έγγραφο της συμφωνίας. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι αυτή η συμφωνία ισχύει όσο η Δανία είναι μέλος της Σέγγεν. Γιατί η συμμετοχή της εξαρτάται κατά κάποιο τρόπο από το Σέγγεν. Υπάρχει λοιπόν ένα εδάφιο, το υπαριθμό 18, το οποίο ρητά αναφέρει πως ε, η συμφωνία ισχύει υπό την αίρεση της συμμετοχής της Δανίας στη συμφωνία Σέγγεν, αλλά δεν βλέπουμε κανένα λόγο η Δανία να εγκαταλείψει το χώρο Σέγγεν στο εγγύς μέλλον. Με αυτά τα σύντομα σχόλια καλωσορίζουμε τη συμφωνία και την ε, θετική διάθεση που έδειξε το Κοινοβούλιο στην επιταχύνη της διαδικασίας για να υπογραφεί η συμφωνία πριν από τη θέση ενισχύ του κανονισμού Eurojust στις 12 Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Περίμενα και εγώ να ακούσω αν θα μας αναφέρετε στην ομάδα και τη συνεργασία. Ξέρετε πως το Κοινοβούλιο αφιερώνει πολύ χρόνο για τη Europol, για τη Eurojust, για το, η Δανία, αλλά δεν το συγκαταλέγεται στην ομάδα. Α, κοινοβούλιο είναι. Έπρεπε να το αναφέρω και αυτό. Γιατί στην υπέροχη αυτή ομάδα δεν ξέρω αν βλέπετε τη συμμετοχή του Συμβουλίου ή την Προεδρία, αλλά το κοινοβούλιο θα μπορούσατε να το αναφέρετε. Ξέρετε, έχουμε κάνει άπειρε συνεδριάσει. Έτσι, μια μικρή υπόδειξη, αν μου επιτρέπετε, την επόμενη φορά που θα αναφερθείτε σε μια ομάδα. Ε, βάλτε το και στο κειμενάκι σα. Άλλωστε, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο ο σχεδιασμό του κειμένου. Είναι και στην πράξη. ότι κάνουμε σήμερα, το θα κάνουμε στην Ολομέλεια. Αυτά μετράνε. Εκτό και αν το κοινοβούλιο δεν έχει την ίδια αξία. Δεν ξέρω αν ε, υπάρχει κάποιο άλλο να μιλήσει πλην των δανών εκπροσώπων. Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δανίας, Περνίλ Μπράινχολτς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ξεκινώντας θέλω ε, εκ μέρους της Δανίας, της κυβέρνησης της Δανίας, να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Να, είδατε τι έξυπνοι που είναι. Αμέσω πρώτο έβαλε το Κοινοβούλιο. Να, σα μάθουμε και τρόπου. Η Δανία θα σα το διδάξει αυτό. Να συνεχίσω λοιπόν. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σα που μα υποδέχεται σήμερα εδώ και που μας επιτρέπει να συστήσουμε το θέμα αυτό κατεπηγόντως τη συμμετοχή στη Eurojust. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες, είναι πολύ σημαντικό για μας, ώστε να μην υπάρξουν λειτουργικές χάσματα σε σχέση με τη λειτουργική συμμετοχή μας ε, στη Eurojust. Όπως ανέφερε και ο πρόσωπος της Eurojust, ε, συμμετέχουμε στη Eurojust από τη θέσπιση της το 2002. Με πολύ στενή συνεργασία στα λιγότερο αλλά και τα περισσότερα περισσότερο γνωστά ζητήματα που έχουν προκύψει ε, σε δίωξη διαφορών δικτύων παρανομίας και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι ζητήσαμε από το Συμβούλιο την άδεια να συνεχίσουμε τη δουλειά αυτή και μετά τις 12 Δεκεμβρίου. Είμαι θα ευγνώμονε που το Συμβούλιο και η Επιτροπή έκαναν δεκτό το αίτημα και που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε σκόπιμο να φέρει το θέμα. Βλέπετε, λέει ο κύριο Μωρέ. Να, να τρόποι Ακούστηκε ήδη ότι η Eurojust ακολουθεί το ίδιο μοντέλο με τη Europol. Και στηρίζεται στο γεγονό στηριζόμενη στο γεγονός ότι είναι κράτος μέλος ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχει και στη Σέγγεν, η Δανία ε, αναγνωρίζεται ότι μπορεί να συμμετέχει Βέβαια η ενδεχόμενη αποχώρηση ή η η αποχώρηση από τη Σέγγεν ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Δανία θα έθετε τέρμα και στη συμμετοχή τη στη Eurojust όπως άλλωστε και στη Europol. Ένα ζήτημα επίση που θέλω να τονίσω είναι ο έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την εκτέλεση, υλοποίηση τη συμφωνία. Και επίση αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με τρίτες χώρε ότι συμμετέχουμε και στον προπολογισμό τη Eurojust. Για μας λοιπόν είναι ευτυχές το αποτέλεσμα η έκβαση αυτής της ε, συνεργασίας και η σημασία της ε, συμφωνίας υψηλή. Περιώνω λοιπόν εδώ την, την ε, παρέμβασή μου. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ και θα ακούσουμε την κυρία Σίπελ και τον κύριο Πίτερσον. Η κυρία Σίπελ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πάντα μου άρεσε η δουλειά σα. Αυτές τι τελευταίε δύο εβδομάδε όμως κάτι έχετε αλλάξει και μου αρέσετε ακόμα πιο πολύ. Μα όχι, απλά λέει ο πρόεδρος, ε, μου αρέσουν κάποιοι στην Επιτροπή και πώς συμπεριφέρονται όταν αντιμετωπίζουν πίεση από το Συμβούλιο. Εγώ όχι, τίποτα δεν άλλαξα. Απλά η ελαζονία του Συμβουλίου μου προκαλεί έκπληξη, τι να πω, και ανικανότητα. Ναι, λέει η κυρία Σίπελα. Να το σκεφτούμε. Καταρχά, είναι πολύ θετικό που όλοι είναι εύτυχοι και ικανοποιημένοι. Συγχαρητήρια ακούμε για την πρώτη αυτή διαδικασία. Αυτό είναι θετικό. Σα ευχαριστούμε. Μα λέει η Δανία. Αλλά κοιτώντα το τι συζητάμε, δεν έχω διάθεση να συγχαρώ για πολλά πράγματα πέρα από το χρονοδιάγραμμα, αλλά κανονικά δεν μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Και δεν θέλω να ακούω και ευχαριστίε. γιατί δεν το απευθύνω αυτό ω ε, κριτική στη Δανία, μάλλον ω κριτική προ όλα τα κρατημέλη. Το λέω ότι επιτέλους θα πρέπει να μάθουν, επιτέλους να παίρνουν πιο πολύ στα σοβαρά τη συμμετοχή τους και την ε, θέση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά ήταν απαραίτητα ε, γιατί πολύ απλά η Δανία ξαφνικά δεν είναι μέλος της Eurojust για κάποιο απίθανο λόγο. Και συγγνώμη που το λέω Κλοντ, αλλά αυτές είναι οι τραχικές εμπειρίες που έχουμε στο opt-out. Όταν κάποιο συμμετέχει σε μια λάσχη, θα πρέπει να σέβεται όλους τους κανόνες της λάσχης. Δεν θέλουμε να ανοίξουμε την πόρτα και τα παραθυράκια για διάφορες διάφορε αποκλήσει από του κανόνε. Αυτό είναι μια γενική προσέγγιση. Σήμερα αφορά την Δανία. Γενικά όμω το λέω και να κάνω και μια άλλη γενική παρατήρηση για το Σέγγεν. Γιατί όπω είπε κάποιο, όσο δεν φεύγει η Δανία από την ζώνη Σέγγεν, εγώ να το θέσω σε πιο διαφορετικό επίπεδο, με κοινικό τρόπο. Έχουμε ακόμα Σέγγεν με όλου αυτού του ελέγχου Αναρωτιέμαι, διαρωτώ με κατά πόσον υπάρχει καν η ζώνη Σέγγεν. Αυτό είναι πολιτική δήλωση και λυπάμαι γι' αυτό και λυπάμαι. Επίσης, γιατί σε λίγα λεπτά θα χρειαστεί να φύγω, γιατί έχω μια άλλη σημαντική ανταλλαγή απόψεων για τα ηλεκτρονικά τεκμήρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Ζίπελ. Το ίδιο λέτε που λέω και εγώ στην Europol. Έχω δαπανίσει ώρες και ώρες εργασίας και η Δανείοι ήταν ευτυχής που άμα περισσώσαμε την κατάσταση αυτή και μαζέψαμε τα σπασμένα. Στο JPSC για παράδειγμα. Το ξέρω γιατί έχω ταμπανίσει πραγματικά ώρες επί ωρών. Αυτά όλα θα πρέπει να είναι κατανοητά και αυτονόητα. Γιατί η Eurojust τα πράγματα τώρα είναι λίγο διαφορετικά. Οι υποδομέ είναι λίγο διαφορετικέ. Θα τεθεί όμω άλλο ένα θέμα στο οποίο θα εμπλέκεται το Κοινοβούλιο. Και αποφασίστηκε αρχικά να μην γίνει η διαδικασία αυτή μέσα στη θητεία, γιατί είχαμε υπερβολικό φόρτο εργασία. Στην πορεία άλλαξε αυτό. Να πω στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο και στην Προεδρία να το έχουν αυτό υπόψη. Οι συντονιστέ λοιπόν δεν ήταν δεδεθμένοι να κάνουν την εργασία αυτή. Αλλά λίγο πριν το τέλο, χτε ψηφίσαμε τελικά. Και θα είχαμε τη συζήτηση. Να το εκτιμήσουμε λοιπόν αυτό. Κύριε Πίτερσον, Ξέρω ότι είσαστε αισιόδοξο άνθρωπο. Να ξεκινήσω ευχαριστώντα εσά, κύριε Πρόεδρε, και όλου του συναδέλφου που επέδειξαν ευελιξία και πνεύμα βοήθειας προς την ε, Δανία σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Παρά το γεγονό ότι σε προσωπικό επίπεδο συμφωνώ λίγο πολύ με όλα αυτά που δήλωσε η κυρία Σίπελ και ζητώ μάλλον λυπάμαι για αυτό το δανέζικο opt το οποίο δημιουργεί θέματα επιθεμάτων διαρκώς. Θα ήθελα να υπογραμμίσω όμως εκ παραλλήλου σε πιο προσωπικό επίπεδο πόσο ευγνώμονες είμαστε πολύ εξημών. Για την ευελιξία που επιδεικνύει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής. Ευχαριστώ λοιπόν για την ηγεσία που επιδείξατε κύριε Μωράης. Να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους εδώ στο Κοινοβούλιο που επέτρεψαν αυτή την ε, γοργή διαδικασία και ουσιαστικά επέλυσαν ένα πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα για την Δανία. Ναι, θέλω το Κοινοβούλιο να χαίρει σεβασμού και να είναι ορατό, να προβάλλεται λέει ο πρόεδρο, όχι να μαζέψω συγχαρητήρια. Να αναγνωρίζει τη βοήθειά του από πλευρά του Συμβουλίου ενίοτε. Αυτό θέλω να τονίσω. Μάλιστα. Άλλο τίποτε. Το Κοινοβούλιο τώρα. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Λίμπε στι 8 και μετά στην Ολομέλεια στη δεύτερη Ολομέλεια του Απριλίου. Και αυτά θα επιλύσουν τα προβλήματά σα. και τεθούν άλλα θέματα όπως ε, με τη Europol, έλατε να μου το πείτε. Ή εμένα ή σε οποιονδήποτε είναι ο διάδοχός μου. Σας ευχαριστώ όλους σας. Και σημειώσαμε τα όσα μας είπατε για τα σχέδια. Ευχαριστούμε τους Δανούς συναντέλφου. Μη σας ε, σοκάρει είναι μου τρόποι. Είναι που είναι το τέλος της θητείας. Θα χειροτρέψουν κι άλλο τα πράγματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι.

Okay, um, colleagues, we've got points 16, 17, 18. Λοιπόν, να δούμε τα σημεία 16, 17 και 18. Ο κύριος Κοράου, εισηγητής, είναι εδώ. Πρόκειται για τη σύναψη πρωτοκόλων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, Δανίας, Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λίθεστάιν και έχει αποφασιστεί από τους συντονιστές να ακολουθήσουμε μια επιτυχημένη διαδικασία στα αγγλικά μόνο και από ό,τι φαίνεται όμως ε, υπό τη θητή αυτή θα ασχοληθούμε μόνο με το πρωτόκολλο της Δανίας ε, καθώς αυτό έχει μόνο ε, γι' αυτό μόνο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφή από το Συμβούλιο. Για τα άλλα πρωτόκολλα μπορούμε να κάνουμε μόνο προπαρασκευαστικά βήματα και το επόμενο Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασχοληθεί με το κύριο μέρος της διαδικασίας συνένεσης. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Κορά, ο οποίος θα παρουσιάσει ε, τις συστάσεις του και για τα τρία πρωτόκολλα. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Η αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac επέτρεψε ε, να έχουν πρόσβαση οι διοκτικές αρχές σε αυτή τη βάση δεδομένων προκειμένου να ερευνούν ε, κύματα τρομοκρατίας και άλλα σοβαρά δικήματα. Ε, θα μπορέσουν οι αστυνομικές αρχές και οι άλλες αρχές επιβολής ε, του νόμου που θα έχουν ε, ειδική άδεια να έχουν πρόσβαση στα εκτελικά αποτυπώματα της Eurodac προκειμένου να μπορέσουν να βρουν την ταυτότητα ή να έχουν τις κατάλληλες προφορίες για να προλάβουν ή να προβούν σε έρευνα για δικήματα τρομοκρατίας ή άλλα σοβαρά δικήματα. Από το 2001 συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δανία, τη Ισλανδία, την Νορβηγία και την Ελβετία για να καθοριστεί το αρμόδιο κράτος για το αίτημα εξέταση φορά και την εφαρμογή ε, των σχετικών ε, τμήματων της Eurodac. Ε, όμως μέχρι τώρα δεν έχει ρυθμιστεί από αυτή τη συμφωνία το θέμα των διοκτικών αρχών. Έτσι λοιπόν τώρα θα πρέπει να προσθεθεί ένα πρωτόκολλο στη Συμφωνία του 2001 για να εισαχθεί η διαδικασία σύγκριση και διαβίβαση των στοιχείων ε, για ε, λόγους επιβολής ε, του νόμου και έτσι οι διοκτικές αρχές θα μπορέσουν να ζητήσουν τη σύγκριση των δεδομένων και των δακτυλικών αποτιμημάτων που έχουν εισαχθεί από τα άλλα συμμετέχοντα κράτη στη Eurodac και στην περίπτωση που είναι απαραίτητο να ε, βρουν να ξεκριβώσουν την ταυτότητα, να λάβουν περαιτέρω πληροφορίε σχετικά με ένα ύποπτο άτομο για σοβαρό έγκλημα ή τρομοκρατία σχετικά με το θύμα. Επίση, η Δανία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία θα βάλουν στη Eurotax σχετικά δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων και μέσω αυτή τη συμφωνία τα δεδομένα αυτά θα μπορέσουν να είναι αντικείμενο ε, διαβούλευση για του ίδιου σκοπού. Το Κοινοβούλιο καλείται να εγκρίνει τη συμφωνία προκειμένου το Συμβούλιο να μπορέσει να την εγκρίνει εξ ονόματο της Ένωσης. Είμαι πεπισμένο ε, ότι θα δώσει το Κοινοβούλιο την έγκρισή του. Παρ' όλα αυτά, βάσει των πληροφοριών που φτάνουν ε, στο Συμβούλιο, θα μπορέσει το Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του μόνο για τη συμφωνία με τη Δανία. Είναι ένα ε, μοναδικό φακελό για τον οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έτσι λοιπόν διαιρεί το φάκελος αυτός από τους άλλους και εγκρίνεται σε αυτή τη θητεία. Στις 11 Απριλίου προβλέπεται να ψηφίσουμε στη Λίμπε και στην Ολομέλεια στη δεύτερη σύνοδο του Απριλίου. Οι συνάδελφοι μπορούν να καταθέσουν ε, τροπολογίες μέχρι τις 8 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοράου. Υπάρχουν σχόλια. Ζεράρ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είμαι Σκιώδης από τους Φιλελευθέρους και θα είμαι σύντομος. Ο εισηγητής μας εξήγησε περί τίνος πρόκειται και συμφωνεί απόλυτα η ομάδα μου με τη θέση που ηθητή και που μας ζήτησε να υποστηρίξουμε. Αυτό ήθελα να πω εγώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Κοράου. Έχουμε λοιπόν στις 8 Απριλίου, στις 12 ε, την κατάθεση τροπολογιών, 11 Απριλίου θα ψηφίσουμε και Απρίλιος 2. Λέμε πάντα, δεν υπάρχει και άλλη επιλογή, έτσι δεν είναι. Έχουμε λοιπόν κάτι στην τελευταία ολομέλεια. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα διακόψουμε για πέντε λεπτά, γιατί έρχεται ο κύριος Νίντερ Μίλλερ για το επόμενο σημείο. σε σχέση με την Σερβία και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Εκτοφυλακής. και 10. 4 και 10 θα ξαναξεκινήσουμε. Peter, we were just pausing for five minutes to wait for you, but you... για πέντε λεπτά για να σε περιμένουμε, αλλά κάτσε και θα ξεκινήσουμε σε δύο λεπτά. Περιμένουμε και κάποιον άλλο. No. She won't be here till 4.30. Could we maybe call her a bit earlier? Maybe we just call her and then we could start with Mr. Niedermüller. massive favour? Yes. Could you think there's a new bottle of red water, you know, yes, fizzy? Could you mind? Thank you. Peter, you would you mind start, starting now? Would you, no, do you mind starting on your point? Is it... Peter, μπορείς να ξεκινήσεις. It's, it's web streamed. Everyone sits there in their offices. Γιατί αναμεταδίδεται και μέσω διαδικτύου. Όλοι κάθονται στα γραφεία και εργάζονται σκληρά, αλλά ακολουθούν φυσικά και την, παρακολουθούν και την επιτροπή μας. Έτσι λοιπόν, ε, το επόμενο σημείο διάταξη είναι υπογραφή συμφωνία περί μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία Σερβία με την κοινή δράση που εκτελείται από Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ξηροφύλαξη Εκτοφυλακή και στη Βοσνία Τζεκοβίνη και στο Μαυροβούνιο. Υπάρχει δυνατότητα συνεργασία. Η Συμφωνία Περικαθεστώτηση είναι να παρέχει ένα νομικό καθεστώ για τι επιχειρήσει του οργανισμού με τα μέλη της ομάδας με εκτελεστικές αρμοδιότητες να μπορούν να αναπτυχθούν στην επικράτεια τρίτη χώρας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Νίντερ Μίλλερ που είναι εισηγητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η ολοκλήρωση συμφωνιών έχει, τέτοιου τύπου έχει ιδιαίτερη σημασία για την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας ε, με τρίτες χώρες, αλλά και για να εξασφαλιστεί ένα σαφές πλαίσιο συνεργασίας με τις τρίτες χώρες για τη διαχείριση των εξωτερικών συνορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, για αυτές τις τρεις συμφωνίες θέλω να υπογραμμίσω κάποιες ουσιαστικέ διαφορές στην, ε, στις διατάξεις που προβλέπουν αυτές. Καταρχάς, διάταξη η οποία προβλέπει πως δεν θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ε, ποινικέ διαδικασίες προβλέπεται μόνο σε μία από αυτές τις τρεις. Επίσης διαφορετική διατύπωση υπάρχει ως προς τα εξαιρετικά δικαιώματα των μελών του συστήματος ε, να αναλάβουν δράση εκ μέρους της τρίτης χώρας και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αβεβαιότητα. Τρίτον επίσης η διατύπωση της ρήτρα για τις εκκρίσεις ε, δεν είναι, ταυτός, δεν είναι απόλυτα ίδια. Ε, τέταρτον, σε σχέση με την ποινική ευθύνη, τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ευθύνη ε, για λόγους υπηρεσιακούς ή τη διάπραξη ενό αδικήματο κατά τη διάρκεια τη εκτέλεση των καθηκόντων πάλι δεν είναι σαφή. Επίση, ε, η διαπραξη σε ποινικέ διαδικασίε ε, δημιουργεί δικαθηκόντων παλι και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία θα πρέπει να ενημερώσουν το χέτερο δυνατό στο το Κοινοβούλιο κατά τρόπο ουσιαστικό για όποια δυσκολία ή αποκλήσεις έχουν εντοπίσει λόγω αυτών των διαφορών. Όταν ε, έχουμε δε στο μέλλον αντίστοιχε ε, διαπραγματεύσεις. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια πλήρη αξιολόγηση πρώτα της τρίτης αυτής χώρας για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μετά μόνο να ξεκινήσει τις συνομιλίες, ενημερώνοντας βέβαια και για το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Για τη διαφάνεια, για να μπορεί το Κοινοβούλιο να αξιολογεί ουσιαστικά τις συμφωνίες αυτές, πρέπει η Επιτροπή να διαθέτει στο Κοινοβούλιο όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα ώστε αυτό να ε, υλοποιήσει, να επιτελέσει το έργο που θεσμικά του ανήκει. Λυπούμε λοιπόν, ιδιαίτερω που το Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να υιοθετήσει αυτές τις συμφωνίες. Μια και το Συμβούλιο δεν έχει ζητήσει τη συνένωση του Κοινοβουλίου ακόμη. Ωστόσο, αυτές οι συμφωνίες είναι αντίστοιχε με αυτές που έχει προβλέψει στο ανακοινωθέν της Επιτροπή. Και έτσι καλό το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει το, το κείμενο αυτό. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ μπορεί να υιοθετήσει σήμερα το κείμενο της, του νέου κανονισμού Σέγγεν και έτσι οι συμφωνίες μπορούν να υιοθετηθούν από το προσεχές Κοινοβούλιο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να λησμονούμε πως η διαχείριση τη μετανάστευση, όπω αναφέρεται, έχει μια ακόμη πολύ σημαντική ε, διάσταση, ένα εργαλείο πολύ σημαντικό που είναι ένα καλώς λειτουργούν σύστημα για το άσυλο. Τρία χρόνια έχουν περάσει και δεν έχει γίνει τίποτα λόγω της τάσης που υιοθετούν στο Συμβούλιο Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών. Λυπούμε που η στενομυαλιά των μελών του Συμβουλίου δεν έχει επιτρέψει την ανάπτυξη της ε, υπηρεσίας για το άσυλο και την ανθεώρηση του Δουβλίνου ικανοποιητικά. Γι' αυτό καλό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει υπηρεσίες που δεν θα περιορίζουν την ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων του ασύλου σε μια διαχειριστική μόνο δραστηριότητα. Ευχαριστώ κυρία Μετσόλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ και θα ήθελα πολύ στο να πω πως το ΕΛΚ υποστηρίζει τον Πρόεδρο στα συμπεράσματά του και τις ε, δηλώσεις ε, για τη συμφωνία με τις βαλκανικές χώρες που θα επιτρέψουν ε, στην Frontex να συμμετέχει σε διάφορες εργασίες ταχεία ανάληψη δράσης για τη Βοσνία Ριζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία με βάση και τον κανονισμό. Ο Τζέραλτ, ο Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ μπορώ να είμαι σύντομο. Υποστηρίζουμε τις συστάσεις ε, του εισηγητού μας. Προσθέτω δε ότι τα συμπεράσματα του τα συμμερίζουμε σε μεγάλο βαθμό. Τα συμμερίζουμε πλήρως. Η Επιτροπή. Oliver Seifert. Πρόεδρε, και εμείς θέλουμε αυτές οι συμφωνίες να τεθούν σε εφαρμογή το χαίτερο δυνατό. Υπάρχει μεγάλη πρόοδος, όπως άλλωστε αναφέρθηκε και σήμερα στη συζήτηση για την ακτοφυλακή και τη Frontex. Ε, οτιδήποτε λοιπόν μπορεί να γίνει από πλευρά των συνομοθετών που θα επιτρέψει την πλήρη θέση εφαρμογή των συμφωνιών είναι για μας ευπρόσδεκτο. Κύριος Νίτερμαϊερ. Όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Άλλο μικρό διάλειμμα. Μέχρι τις 4.30 με την κυρία Ζίπλ, η οποία δεν μπορεί να έρθει πιο νωρίς για το θέμα της.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

Okay, colleagues, um, we'll get started. There's one shadow we're waiting for him to come, but... Ωραία, μπορούμε να ξαναρχίσουμε αγαπητοί συνάδελφοι, περιμένοντα να έρθει και μια ακόμη συνάδελφο. Ολοκληρώνουμε την ε, συνεδρίαση με 7 έγγραφα εργασία, Η κυρία Ζήπελη, συγγήτρια. Δεν θα σας πω τίποτα. Birgit, εσύ. Ευχαριστώ, Κλοντ. Κατόπιν της παρουσίας του πρώτου γράφου εργασίας αρχές ε, Δεκεμβρίου, με τα προηγούμενα έγγραφα Φεβρουάριο και Μάρτιο, μπορώ να σας παρουσιάσω με ικανοποίηση το ένα έγγραφο που έχουμε με το συναφό από τους Πρασίνους, για τα ενδικά μέσα και το άλλο με τον κύριο Γνάσο Κοράου που εξετάζει τη διαδικασία επιβολής και διατήρησης των ε, εντολών δηλαδή διατήρηση των εγγράφων. Για να δούμε λοιπόν τι προβλέπετε σε αυτά που συμφωνήσαμε με το Ρωμαίο Φρανς για τα ενδικά μέσα. Δεν μπορεί ο ίδιος να είναι παρόν σήμερα εδώ. Έχουμε όμως δουλέψει και πάνω στα σχόλια, οπότε μπορώ να μπω σε κάποιες λεπτομέρειες, ξεκινώντας με την κοινοποίηση του θέματος. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι θεμητοί να μην γίνεται κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο για κάποια δεδομένα τουλάχιστον, για κάποιους τύπους δεδομένων. Αλλά οποιοδήποτε, οποιοδήποτε περιορισμός του δικαιώματος κοινοποίησης περιορίζει σημαντικά το δικαίωμα στην ε, υπεράσπιση και άρα στη δίκαιη δίκη. Άρα τέτοιες, ε, τέτοια εντάλματα πρέπει να διέπονται από πολύ αυστηρούς κανόνες και συμπληρωματικές ασφαλιστικές δικλείδες που προτείνουμε εμείς. Τα εκ των προτέρων ε, ένδικα βοηθήματα και όχι μόνο στην πρόταση αυτή αλλά και σε άλλα νομοθετήματα που ισχύουν ήδη δεν καλύπτονται για την ασφάλεια, για την διατήρηση και για την διάδοση των, ή την κοινοποίηση των στοιχείων. Άρα αυτό αποβαίνει βάρος και των κατηγορουμένων αλλά και τρίτων που ενδεχομένω να ε, αφορά το ένταλμα παραγωγής και διατήρησης. Επίσης είμαστε πεπισμένοι ότι η πρόταση πρέπει να ξαναδιατυπωθεί εκεί που γίνεται λόγος για τις αρχές της χώρας ε, όπου αναπτύσσεται η υπόθεση αλλά και της χώρας διαμονές. Για να μην υπάρχει παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ζητούμε να υπάρχει κοινοποίηση των κρατών που εμπλέκονται σε αυτά τα εντάλματα και ενδεχομένως ακόμη και ε, απέτηση για άδεια πριν από την κοινοποίηση, όχι απλή κοινοποίηση δηλαδή. Πριν από την ε, διάθεση των εγγράφων και όχι απλή κοινοποίηση. Επίσης ε, στις κατηγορίες των δεδομένων αλλά και στις ασφαλιστικές ε, δικλίδες. Επίσης για, τις, για τα εκ των υστέρων ενδικά βοηθήματα. Πάλι δεν είμαστε ικανοποιημένοι διότι θεωρούμε ότι η αποτελεσματική αποκατάσταση των δικαιωμάτων δεν εξασφαλίζεται εάν ο ενδιαφερόμενος ενημερωθεί είτε καθόλου είτε ε, σε πολύ ύστερο στάδιο και αν ενημερωθεί μόνο για το κράτος έκδοσης του εντάλματος και το οποίο μπορεί να μην είναι το κράτος διαμονής. Και αν εναπόκειται στο ε, δίκαιο του κράτους του εν λόγω η κάλυψη, η πρόβλεψη των αδικών βοηθημάτων. Άρα δεν μπορεί να αποκατασταθεί ε, στα δικαιώματά του σε περίπτωση που ήταν παράνομη η παραγωγή αυτού του υλικού. Έχει πολύ μεγάλη σημασία βεβαίω να υπάρξει η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και με κανόνες αποκλεισμού αλλά και με κανόνες σε σχέση με την ε, επεξεργασία και την περαιτέρω διοχέτευση των στοιχείων. Αυτό είναι το ένα. Μπορεί επίσης να υπάρξει οικονομική αποζημίωση για, τον, για το υποκείμενο, για τον δικαιούχο ή ιδιαίτερα σε περίπτωση που συστηματικά χρησιμοποιούν οι αρχές έκδοσης ε, αυτές τις μεθόδους. Εδώ επιδιώκουμε και τη δημόσια λογοδοσία σε σχέση με τη χρήση του εγγράφου. Ιδιαίτερα λοιπόν τονίζουμε πως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η Επιτροπή με, το, με την αιτιολογία που προβάλλει ε, παραβλέπει τελείως το δικαίωμα σε ασφάλεια δικαίου, γιατί ούτε ο θεμελιώδης χάρτης, ούτε η Συμφωνία για τα ανθρώπινα δικαιώματα επιτρέπουν ε, την υπαγωγή των δικαιωμάτων αυτών σε άλλα δικαιώματα ή ασφαλιστικές δικλείδες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πέρασω το 7ο έγγραφο εργασία που συντάξαμε στη συνεργασία με τον Ιγνάσιο Κοράου. για την επιβολή των ε, ενταλμάτων. Όταν λοιπόν δεν ανταποκρίνονται οι υπάρχοι των υπηρεσιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει στο εθνικό δίκαιο. Αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε αμφίβολης ποιότητας κίνητρα. Φερρυπίν μπορεί κάποιοι να επιλέξουν να ε, ορίσουν αντίκλητο στο κράτος που έχει τις πιο ευνοϊκές συνθήκες ή μπορεί ένα κράτος να επιλέξει για να γίνει πιο ελκυστικό προς τους παρόχους υπηρεσιών πιο ευνοϊκή νομοθεσία. Άρα χρειάζεται περισσότερο εναρμονισμένο πλέγμα διατάξεων. Και επίσης επισημαίνουμε ότι η προθεσμία για την εκτέλεση των ανταλμάτων, όπως ε, προτείνεται στο σχέδιο του κανονισμού είναι πολύ μικρή, πολύ στενή και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερα πιεστική αλλά γενικά για τους ε, παρόχους ε, υπηρεσιών, είτε θα έχουν τη δυνατότητα να επαληθεύσουν την νομιμότητα των ανταλμάτων Άρα είτε πρέπει να γίνουν χωριστά, χωριστές προβλέψεις ανάλογα του μεγέθους επιχείρησης για τα αντέλματα ή πρέπει η προθεσμία να παραταθεί γενικά. Εν τέλει, στη διαδικασία για επιβολή και τήρηση του άρθρου 14 χρειάζεται επιστολή δουλειά. Πρώτον, γενικά υπάρχουν αμφιβολίες για το αν θα πρέπει ο πάροχος ε, υπηρεσίας να παληθεύει ο ίδιος αν υπάρχουν λόγοι απόρριψης. Επίσης, μπορεί κάποιοι πάροχοι να μπουν στο πειρασμό να ερμηνεύσουν υπερβολικά ευρέως τις διατάξεις αυτές. Και πάλι οι αρχές της χώρας επιβολής και ενδεχομένως και της χώρας ε, διαμονής του εμπλεκομένου πολίτη πρέπει σε πρώιμο στάδιο να συμμετέχουν στη διαδικασία. Είναι πολλά λοιπόν τα ζητήματα που αγείρονται και πολλά εκείνα που είχαν αγερθεί και κατά την παρουσίαση προηγούμενων ε, εγγράφων εργασίας. Διερωτώμεθα λοιπόν πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρία χρόνια μόλις ε, μετά, ε, μετά την ανάληψη αυτού του έργου να παρουσιάζει αυτές τις προτάσεις και πώς μπορεί με όλες τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί από το Κοινοβούλιο, από την Κοινωνία των Πολιτών, από τους ειδικού στα θέματα της προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων, αλλά και από τους παρόχου τους ίδιου, και μην ξεχνάμε και από κάποια μέλη, ε, κράτη-μέλη, να επιμένει να καταθέτει αυτέ τις προτάσεις. Ω εκ τούτου και συμπερασματικά, μπορώ να σα πω ότι δεν αισθάνομαι καθόλου άσχημα αν δεν ολοκληρώσουμε αυτή τη δουλειά εμεί ω Κοινοβούλιο, το δικό μα κομμάτι. Χαίρομαι και είμαι περήφανη που δώσαμε αρκετό χρόνο για να αναλύσουμε ει βάθο την πρόταση. Γιατί μόνο έτσι μπορέσαμε να ε, εντοπίσουμε τι ελλείψεις, τα προβλήματα. Ενώ το Συμβούλιο στόχευσε σε μια επιτυχημένη διαδικασία και δεν κατάφερε να δει τι δυσκολίε ε, των προτάσεων. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ θερμά όλου και εισηγητές ε, τις υπηρεσίες τους, τα γραφεία τους και όλη τη γραμματεία της Επιτροπής μας για την πολύ καλή συνεργασία σε αυτό το σημαντικό θέμα. Είμαι επιπισμένη ότι η δουλειά που έχουμε κάνει όλοι μαζί σε όλα αυτά τα έγγραφα εργασία μας επιτρέπει να έχουμε μια πολύ καλή βάση ώστε σε μεταγενέστερο στάδιο να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Να κάνουμε αυτό δηλαδή που έπρεπε εξ αρχής να έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλύτερη νομοθεσία. Ευχαριστώ. Um, ευχαριστώ. Ο κ. Κράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την συγγητρία την κυρία Σίμπελ, το προσωπικό της και τη γραμματεία της Επιτροπής Λιμπέλ για την εξαιρετική συνεργασία και την υποστήριξη το έγγραφο εργασίας που θα παρουσιάσω αφορά το θέμα της εκτέλεσης της Ευρωπαϊκής Εντολής Υποβολής Στοιχείων και Εντολής Διατήρησης Στοιχείων και συγκεκριμένα την προθεσμία που υπάρχει υπηρεσιών να έχουν για να απαντήσουν στην εντολή της δικαστικής αρχής στη διαδικασία της εκτέλεσης. Ό,τι αφορά τις κυρώσεις, το άρθρο 13 της πρότασης της Κομισιόν αφήνει την ελευθερία στα κράτη-μέλη να προβλέψουν παρεκκλήσεις για χρηματικές κυρώσεις που θα εφαρμοστούν σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση από τους παρόχους υπηρεσίων των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον κανονισμό. Οι κυρώσει θα πρέπει να είναι αναλογικέ και αποτρεπτικέ και πραγματικέ. Βέβαια, εκτιμούμε το γεγονό ότι αφήνεται στα κρατη η δυνατότητα να εφαρμόσουν ποινικέ ή διοικητικέ κυρώσει που να είναι πιο συνεκτικέ με την αντίστοιχη νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά, προκειμένου η διάταξη αυτή να μπορέσει να είναι αποτελεσματική, θεωρώ ότι μία εναρμόνιση των κυρώσεων τουλάχιστον ελάχιστη χρειάζεται. Αν θέλουν να αποφευθούν φαινόμενα forum shopping, θα πρέπει να υπάρχει μία ελάχιστη υποχρέωση για όλα τα κράτη-μέλη. Ε, διαφορετικά, οι παροχοί θα επέλεγαν τα κράτη-μέλη όπου έχουμε χαμηλότερες ποινές. Εξάλλου θα υπήρχε και κίνδυνος να ξεκινήσει ένας ανταγωνισμός προς τα κάτω για τον καθαρισμό των κυρώσεων μεταξύ των κρατών κοιλών έτσι ώστε να προσελκύζουν περισσότερους παρόχους ε, και ε, να προβλέπουν τις ελάχιστες ποινές στην επικρατειά τους. Μία άλλη πτυχή που πρέπει να αξιολογηθεί οπωσδήποτε όταν θα καθοριστούν οι κυρώσεις αφορά τις διαστάσεις των παρόχων. Δεν μπορούμε να βάλουμε στο ίδιο επίπεδο την Google με μία μικρή τοπική startup. Η λύση που βρήκε το Συμβούλιο να μειώσει τις κυριώσεις σε σχέση με την ετήσιο όγκο εργασιών ακολουθεί την ίδια λογική ισότητας που και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναζητήσει. Η σωστή εφαρμογή αυτών των κυρώσεων συνδέεται άρρηκτα με όσα είπα και αποτελεί ε, την συνήθη διαδικασία. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εγγυώνται πάντα ότι ε, ε, συνδυάζονται οι κυρώσεις όπως πρέπει και γίνονται σεβαστές και θα πρέπει να παρακολουθείται η πραγματική εφαρμογή τους. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε φαινόμενα άγρας δικαστηρίου. Ένα άλλο σημείο αφορά τη διαδικασία εκτέλεσης των ευρωπαϊκών εντολών υποβολής και διατήρησης στοιχείων, κυρίως σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα που αφήνεται στον πάροχο να αντιταχθεί στην εκτέλεση βάσει δικής του προσωπικής αξιολόγησης για το αν υφίσταται οι διαδικασίες για την έκδοση και κάτι που με προβληματίζει αφορά τη δυνατότητα ο πάροχος να αντιταχθεί ε, στην ε, έκδοση, αν ε, παραδείγματο χάρη είναι πρόδειλ ε, η εντολή, ε, κατάφορα, συγγνώμη, αν προδήλω παραβιάζει την χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν δίνεται σε έναν ιδιώτη τη δυνατότητα να αξιολογηθεί ένα εντολή συνάδει με το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και επομένω κρίνει το δικαστικό σύστημα του κράτου έκδοση. Νομίζω ε, ότι θα μπορούσε πάντοτε να χρησιμοποιεί τέτοιε δικαιολογίε ο πάροχο σε όσα έχουμε στην πρόταση κανονισμού. Δίνεται ε, η ευθύνη, η ευθύνη πρέπει να δοθεί στο κράτος μέλος ε, όπου βρίσκεται ο πάροχος. Αν τελικά αντιταχθεί ε, ένας πάροχος ε, τόσο ε, περισσότερο θα τον προτιμούν όσοι θέλουν να έχουν μυστικά. Και βέβαια αυτό μπορεί να ευνοήσει και παρόχους υπηρεσιών με περισσότερα μέσα που μπορούν να βασίζονται στην ύπαρξη, υφιστά, στην ύπαρξη νομικών μελετών. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να περιοριστούν οι λόγοι ε, για τους παρόχους, ε, παραδείγματος χάρη, ε, σε πολύ περιοριστικές καταστάσεις ή σε μη δικαστικές καταστάσεις. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κριτήριο που εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία το θέμα της επιστολής και θα είχε ε, κάποια αρνητική συνέπεια, να δώσει στον πάροχο ε, να ε, μπορέσει να κατηγορήσει ένα κράτος μέλος ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό δεν ακολουθεί την υποχρέωση της αμοιβαία αναγνώρισης που πρέπει να βασίζεται η δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσεις και δυστυχώς η Ένωση είναι πολύ μακριά από το να την έχει υλοποιήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και να πάμε στην Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να διαφωνήσω με τον ε, βουλευτή σε ό,τι αφορά την αντίθεση που εκφράζει στην έκφραση, στην ε, άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την τοποθέτηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, το μελετήσαμε με πάρα πολύ καιρό και καταλαβαίνω ότι δεν προκαλούν ε, έντονε αντιθέσεις όλε οι τοποθετήσει, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η άποψη των ε, ατόμων που εργάζονται στον κλάδο και των εμπλεκομένων φορέων και των παροχών ε, υπηρεσιών και είναι κρίμα που στην όλη αυτή τη διαδικασία διαβούλευση δεν συμμετέχει εξίσου το Κοινοβούλιο. Είναι πιο απλό να διαβουλευτούμε με εμπρεγνώμονε των κρατών μελών σε τέτοια ζητήματα. Αλλά θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα ήταν καλό και θα χαρούμε να συζητήσουμε περαιτέρω ε, προτάσεις με το επόμενο κοινοβούλιο βάσει των ε, εγγράφων εργασίας που παρουσιάστηκαν και καταρτίστηκαν και θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε την πρόταση. Σε ό,τι αφορά τα διάφορα θέματα, δεν θα επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά να πω το εξή. Μία από τις βασικές προ... προκλήσεις είναι να βρεθεί μία ισορροπία, να είναι και αποτελεσματικό το εργαλείο και να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα, το να ε, ε, επαναλάβουμε και να δημιουργήσουμε παράλληλους μηχανισμούς με τον EIO και τον υφιστάμενων μηχανισμούς δεν ε, αποτελεί σκοπό μας. Δεν θέλουμε να υπάρχει επικάλυψη σε σχέση με τα υφιστάμενα συστήματα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε την ισορροπία αυτή και αυτό αποτελεί και τη δυσκολία στο φάκελο αυτό. Συζητήσαμε πολλά από τα θέματα τα οποία ακούσαμε σήμερα σε ό,τι αφορά την κοινοποίηση, για παράδειγμα, του υποκειμένου. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έννοια. Και συμφωνούμε ότι το άτομο θα πρέπει να ενημερώνεται προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να ασκεί και τα δικαιώματά του και να αμφισβητήσει την νομιμότητα της διαδικασίας. Όταν πρόκειται για τρίτο άτομο το οποίο δεν είναι υποπτό και κατηγορούμενο για κάποια διαδικασία θα πρέπει να ενημερώνεται σε κάθε περίπτωση. Το θέμα λοιπόν είναι πότε θα πρέπει να γίνεται αυτή η κοινοποίηση. Σε ποια χρονική στιγμή. Στις έρευνες συχνά υπάρχει ανάγκη να διατηρείται το απόρριτο της διεξαγωγή των ερευνών μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Αυτό λέμε λοιπόν στην πρόταση. Και αυτό συνάδει και με την σχετική οδηγία 13.3. έχουμε και διατάξεις που προβλέπουν την πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία. Σε ό,τι αφορά την κοινοποίηση ενός άλλου κρατούς μέλος και αυτό θα μας απασχολήσει θεωρώ και στο μέλλον σε ό,τι αφορά το φάκελο αυτό. Και πάλι να έχουμε υπόψη μας ότι εδώ θα πρέπει να βρούμε λύσεις. Να βρούμε λύσεις οι οποίες δεν θα επιβαρύνουν υπερβολικά το εργαλείο αυτό. θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό το εργαλείο. Αυτή η γενική προσέγγιση εισήγαγε ήδη κάποιες υποχρεώσεις κοινοποίηση και εδώ θα συζητήσουμε περαιτέρω θεωρώ το πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά. Χωρίς να επιβαρύνουμε το εργαλείο, επαναλαμβάνω. Για τα ενδικά μέσα εξάντα, εκ των προτέρων. Οι κατηγορίε επίση δεδομένων αποτελούν μια περαιτέρω κατηγορία, μια, ένα περαιτέρω θέμα το οποίο θα συζητήσουμε επισταμένο στο μέλλον. Δεν θέλω να επισέλθω τώρα σε λεπτομέρειε. Θα συζητήσουμε θέματα όπως οι μεταφορές δεδομένων για να συνάδουν με τις κανόνες για την προστασία των δεδομένων σε ό,τι αφορά λοιπόν τα δικά μέσα ex post εκ των υστερών. Πολύ σημαντικό θέμα και αυτό κατά τη γνώμη μας και νομίζω ότι το άτομο θα πρέπει να γνωρίζει ποιος έχει πρόσβαση στα, δεδομένα του και θα πρέπει να έχει και τα ενδικά μέσα για να ασκήσει τα δικαιώματά του. Να λαμβάνουμε υπόψη όμως το γεγονό ότι λειτουργούμε σε ένα τομέα νομικών συστημάτων και ενδικών συστημάτων με μεγάλε διαφορέ και με μεγάλε αποκλήσει μεταξύ κρατών μελών. Άρα, το επίπεδο εναρμόνιση. Ε, επιλέξαμε να μην εναρμονίσουμε τα ενδικά μέσα αυτά και να αναφέρουμε μόνο την αρχή ότι θα πρέπει να υφίστανται ενδικά μέσα. σε δικαστικές υποθέσεις όπου κάποιος κατηγορείται ή κάποιος είναι ύποπτος ή ένα άτομο τρίτο το οποίο δεν είναι ύποπτος αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να είναι σε θέση να αμφισβητεί την νομιμότητα της διαδικασίας. Αυτό υπερβαίνει αυτά τα οποία προβλέπονται σε κάποια κρατημέλη. Ε, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό μπορεί να σημαίνει οικονομική αποζημίωση. Αξίωση η οικονομική αποζημίωση. Δεν έχουμε της διαδικασια αυτο υπερβαινει αυτα τα οποια προβλεπονται σε καποια κρατημελη σε ορισμενες περιπτωσεις λοιπόν στον βαθμό για να εναρμονίσουμε τα συστήματα αυτά. Σεβόμαστε τις διαφορές και τις αποκλήσει που υπάρχουν μεταξύ εθνικών συστημάτων αποφασίσαμε λοιπόν, το σκεφτήκαμε αυτό στην αρχή, αλλά αποφασίσαμε να μην το πράξουμε ακριβώ επειδή υπάρχει διαφορά στα ενδικά συστήματα των κρατών μελών. Σε κάποια συστήματα, για παράδειγμα, ο δικαστή είναι αυτό ο οποίο αποφασίζει τι γίνεται σε ό,τι αφορά τα τεκμήρια τα, τα οποία προσάγονται στο δικαστήριο, τα αποδεκτικά στοιχεία τα οποία προσάγονται. Ε, ενδεχομένω αυτό να είναι και πιο κατάλληλο να γίνει σε κάποιο άλλο οριζόντιο μέσο. Το οποίο ενδεχομένω να υποβάλει ω πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον. Και τώρα να δώσω το λόγο στη συναδελφό μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ για τα έγγραφα εργασία αυτά που μα δείξατε, που μα δώσατε. Θέλουμε να συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειε κάποια από τα στοιχεία που θέσατε, αλλά να σας δώσουμε και κάποιε πρώτε πρώτες Εργαζόμαστε σε ένα σύστημα όπου μόνο το 1% των κυβερνοεγκλημάτων α, εκδικάζεται τελικά. Γιατί στις πιο πολλές περιπτώσεις τα αποδεκτικά στοιχεία έχουν ήδη διαγραφεί όταν ξεκινάει η έρευνα. Δεν υπάρχει σύστημα αρχιοθέτηση των ε, αποδεκτικών στοιχείων και οι τρέχουσες διαδικασίες έχουν ως αποτέλεσμα να προσάγονται τα αποδεκτικά αυτά στοιχεία, αλλά να, να μην χρησιμοποιούνται και να μην περνάμε ποτέ στο τέταρτο και τρίτο και τέταρτο μάλλον επίπεδο ε, ε, έρευνα. Μόνο 4% των περιπτώσεων κατάχρησης. Οι πλάνησες αναλύκων τελικά εκδικάζονται. Εκτιμούμε τις μεθόδους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απλά δεν έχουν αποδεκτεί ε, επαρκή σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά αυτά αποδεκτικά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τώρα την συμμετοχή των ε, κρατών μελών, εξάντε ή εξπόστε. Ο λόγος τον οποίο επιλέξαμε να αυξήσουμε τους ελέγχους στο, στη χώρα έκδοσης και όχι να γίνεται δεύτερος έλεγχος στο ε, κράτος αποδοχής είναι ότι διαπιστώσαμε ότι το δεύτερο κράτος μέλος ουσιαστικά δεν έχει πολλά να προσθέσει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του ατόμου που είναι υπό έρευνα. Γιατί ουσιαστικά το κράτος υποδοχής δεν έχει πληροφορίες για το άτομο το οποίο είναι υπό έρευνα. Γιατί οι υπηρεσίε αυτές ουσιαστικά ε, χορηγούνται παγκοσμίω ε, από μια διεθνή βάση δεδομένων. Έχουμε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι πληροφορίες σε 93% των περιπτώσεων ο στόχος ε, ερευνών είναι οι αρχέ ε, ερευνών. Σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες, συμφωνούμε ότι είναι πολύ φιλοδόξες. Και αυτό έχει να κάνει με τις ανάγκες που έχουμε και με το γεγονός ότι δεν έχουμε σύστημα αρχιεφέτησης των, των τεκμηρίων των αποδεκτικών στοιχείων. Αν δεν, δεν μπορούμε λοιπόν να ε, έχουμε εντάλματα για να παγώνουν τα στοιχεία αυτά, αν δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία, πολύ απλά θα διαγράφονται τα στοιχεία σε ό,τι αφορά την σύγκριση μιας τοπικής ε, νεοφιλελευθερία και τη Google. Προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη τι διαφορέ μεταξύ των διαφόρων παρόχων υπηρεσιών και μα ανησυχεί το γεγονό ότι ε, δεν καλύπτονται καν από τον κανονισμό μα ε, κάποιε τοπικέ επιχειρήσει οι οποίε δεν λειτουργούν σε διασυνοριακό επίπεδο. Μόνο όταν λειτουργήσουν σε διασυνοριακό επίπεδο ουσιαστικά εμπίπτουν στον πεδίο και προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη και τι διαφορέ που προκύπτουν από τα διαφορετικά μεγέθη ε, επιχειρήσεων. Θα θέλαμε να υπάρχει μια αμοιβαία αναγνώριση, ένα σύστημα αμοιβαία αναγνώριση. Αυτό ουσιαστικά προσπαθούμε να πετύχουμε. Να δημιουργήσουμε ένα σύστημα όπου ο ρόλο του κράτου θα περιορίζεται στι περιπτώσει εκείνες όπου δεν μπορεί να υπάρχει άμεση συμμόρφωση και ο πάροχο υπηρεσία θα έχει πολύ περιορισμένα δικαιώματα να αρνηθεί, αλλά για προφανή ζητήματα. Δεν μπορούμε λοιπόν να τους δώσουμε οποιαδήποτε ουσιαστική αρμοδιότητα ελέγχου. Αν χρειαστεί λοιπόν να εφαρμογή, αυτό προϋποθέτει ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο στο άλλο κράτος μέλος. Σοφή, θέλετε να πάρετε το λόγο να σχολιάσετε, κυρία Ντφέλτ. Όχι, μάλιστα. Σχόλια εκτό μικροφώνου. σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Έχουμε ένα ψήφισμα του 2017 του έγκλημα, το οποίο μας καλεί να υποβάλουμε τέτοιες προτάσεις και απαριθμεί μια σειρά κριτηρίων τα οποία θα πρέπει να σεβαστεί η πρότασή μας. Τα πήραμε πάρα πολύ σοβαρά αυτά που μας είπατε τότε και θα τα βρείτε λοιπόν τα κριτηρία αυτά στην πρότασή μας. Μας εκπλήσει το γεγονό ότι τώρα έχετε διαφορετική προσέγγιση. Προσβλέπουμε φυσικά στη συζήτηση και προσβλέπουμε και στη μελλοντική συνεργασία με το επόμενο κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τις δύο. Ιργίτ και κύριε Κορά. θέλετε να απαντήσετε. Πολύ σύντομα, γιατί εξεπλάγει από όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Όταν συζητήσαμε επί του εγγράφου μας και κάτι παρόμοιο έκανε το Συμβούλιο και μιλήσαμε για την εμπλοκή δεύτερου τρίτου κράτου μέλου. Ποτέ δεν είπαμε στο γραφείο μα ότι αυτό πρέπει να γίνει από την πρώτη στιγμή που ξεκινάει η έρευνα, αλλά νομίζω πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι ή πιο ακριβεί για να δούμε ποιο είναι η κατάλληλη στιγμή να εμπλακεί ένα κράτο μέλο, κυρίω όταν ένα άτομο δεν είναι στο κράτο μέλο έκδοση ή ίσω ε, ούτε καν στο κράτος που βρίσκονται τα δεδομένα και για το 93%. Καταρχήν, αν μιλάτε για 93%, εξακολουθούμε να έχουμε 7% όπου οι άνθρωποι και το έγκλημα δεν είναι στο ίδιο κράτο μέλο και θα θέλαμε και πάλι να ελέγξουμε. Αυτό ο αριθμό προέρχεται από μια συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων και δεν ταιριάζει με όλα τι κατηγορίε δεδομένων που έχουμε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ ακριβεί για όλε αυτέ τι ερωτήσει. Και για το ψήφισμα, συγγνώμη, αυτό είναι κάτι που αφορά την αρχική Επιτροπή των ερχών. Συμφωνούμε πολύ γρήγορα, όλοι θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή και πρέπει να το σκεφτούμε. Όμως ε, θα πρέπει να πούμε περισσότερο σε λεπτομέρειες. Και λυπάμαι που ακούω τις συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο, ότι καταρχήν προσπαθούν να επανεφεύρουν τη διατήρηση. Δεν είναι καλό αυτό. Και δεύτερον, καθυστερούν πάρα πολλέ συζητήσει. Μάλιστα, τώρα μιλάνε και για κακοποίηση παιδιών. Έχουμε νομοθεσία για κακοποίηση παιδιών. Δεν ξέρω γιατί πράγμα μιλάμε εδώ. Α είμαστε λοιπόν πιο συγκεκριμένοι. Α πάρουμε τα πράγματα σοβαρά. Χαίρομαι που ακούω την Κομισιόν ήδη υιοθέτησε μία-δύο ιδέες από το Συμβούλιο και μπορώ να ελπίσω ότι μπορεί να ισχύσει το ίδιο και για ιδέες του Κοινοβουλίου. Γιατί πρέπει να είμαστε ταχεί σε αυτούς τους τομείς, αλλά το να είμαστε ταχεί δεν είναι το μόνο που πρέπει να διασφαλίσουμε. Όπως είπα, πρέπει να κάνουμε και καλύτερη νομοθεσία και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα είναι ένα ακόμη νομοθέτημα που θα καταλήξει ενώπιον ενός δικαστηρίου. Έτσι λοιπόν ε, έχει νόημα να ελέγξουμε τα πάντα και στα δύο αυτά έγγραφα εργασία ε, που αναφέρουμε σήμερα δεν είναι το μόνο, αλλά ε, έχουμε ενώπιόν μας τι γίνεται και με τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, μπορεί να αποτελεί και ένα μοντέλο για διεθνή συμφωνία και άλλες διεθνείς συμφωνίες επίσης μπορεί να προκύψουν από αυτό. Νομίζω ότι έχει νόημα να εργαστούμε σωστά έτσι ώστε να έχουμε ένα καλό παράδειγμα που θα μπορούσαμε να εκπονήσουμε περαιτέρω. Και ναι, ανυπομονώ για την καλή συνεργασία, για περαιτέρω καλή συνεργασία, όχι μόνο με τους συναδέλφους εδώ στο Κοινοβούλιο, με αυτούς που είναι τώρα, με αυτούς που μπορεί να επανέλθουν για την επόμενη θητεία και περαιτέρω συνεργασία με το Συμβούλιο, με την Κομισιόν, έτσι ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον στην επόμενη Προεδρία να έχουμε μια αποτελεσματική πρόταση και που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις ανησυχίες και όπου θα βρούμε μία λύση προκειμένου να μην ε, έχουμε μία ακόμη εντολή έρευνας αλλά να έχουμε κάτι αποτελεσματικό. Ίσως αν όχι για όλα τα δικήματα, αλλά για πιο συγκεκριμένα πράγματα που συζητάμε και έχουμε επιτάπητος. Ο κύριος Κοράου, όχι. Ευχαριστώ, Μπριγκίτ, ευχαριστώ και την Κομισιόν. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και στην επόμενη θητεία. Αυτό ήταν το τελευταίο σημείο. Έχουμε και μια συνάντηση αύριο στις 8.30 το πρωί και η επόμενη συνεδρίασή μας θα είναι περαιτέρω τον Απρίλιο.